Ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο η συζήτησή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή, όλους όσοι παρέμειναν στην αίθουσα. Συνεχίζεται αύριο συνεδρίαση από τις 9 η ώρα το πρωί. Έχετε την ημερήσια διάταξη που είναι διαθέσιμη και στην επίσημη στο σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και όλους όσους εργάζονται στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που μείνανε μαζί μας μέχρι τόσο αργά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ.